τα πρακτικά των συνεδριάσεων από 28 και 29 Μαρτίου και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί υπάρχουν. Υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς αυτά. Όχι, από ό,τι βλέπω, άρα λοιπόν τα πρακτικά εγκρίνονται. Ο κύριος Δήμητας Στογιάννοφ έκανε μια πρόταση από 8 Νοεμβρίου 2000.